Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Καταρχήν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Τα πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα ε, είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Δεν βλέπω. Έχει κάποιος αντίρρηση. Όχι. Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Περνάμε στο πρώτο σημείο της μερίσιας διάταξης για σήμερα. Δήλωση της Αντιπροέδρου